Good morning, everyone. I would uh, propose you to slowly start the meeting today. Καλημέρα σας. Ας αρχίσουμε, παρακαλώ. Okay. I want to introduce the first point on our agenda. Το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη να πούμε χρόνια πολλά στον Πολ Μπράνον. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες πέμπτη πρωί, το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Χωρίς καμία άλλη τροποποίηση εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Αν συμφωνείτε, ορισμένες ανακοινώσεις σε σχέση με το πρόγραμμα υποστήριξης της μεταρρύθμισης, επειδή υπάρχει μεγάλο φόρτος εργασίας στο τέλος της θητείας, οι συντονιστές ε, πρότειναν να μην γίνει καμία πρόταση, πρόταση γνωμοδότησης και οι τροπολογίες θα ενταχθούν από την Πρόεδρο. Η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι 16 Οκτωβρίου στις 11 και ελπίζουμε να ε, μπορέσουμε να ψηφίσουμε τον Νοέμβριο. Μετά έχουμε ένα workshop για τις ε, στεφανίες νόσους από τον Καπεσόν Ρουής 9 ε, Οκτωβρίου από τις 10 δεν έχουμε ακόμα αίθουσα, σας καλούμε να παρευρεθείτε. Σήμερα έχουμε 19 γλώσσες και όπως ξέρετε έχετε τον φάκελο και ηλεκτρονικά και θα γίνει απευθείας μετάδοση. Προτείνω λοιπόν το πρώτο θέμα σήμερα, η εφαρμογή του Euro 5 για την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων και τετρακύκλων. 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14 και 15 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. The vote is closed. Εγκρίνεται. Ένα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δύο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5 και 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική άρχεται. It's Πέρας. Εγκρίνεται. Now Ψηφίζουμε τώρα για τις τροπολογίες για τη σύσταση της διευκόλυνσης συνδέοντας στην Ευρώπη. Τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. The vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Εγκρίνεται, με συγχωρείτε. 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά έλεγχος. And Πέρας. Εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές έλεγχος πέρας εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, απόχέ, απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά, απόχέ, απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά, απόχέ. εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, απόχέ. εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται. ΕΛΚ. Δείξτε μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Πέρας. Εγκρίνεται. Now. Τώρα ψηφίζουμε τις τροπολογίες για τη θέσπιση πολιετού σχεδίου για τις αλλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βένθο-πελαγικών αποθεμάτων στη Δυτική Μεσόγειο θάλασσα. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35 υπέρ. Πάλι 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 πρώτο τμήμα υπέρ κατά Ελέγχουμε. 42 πρώτο τμήμα. Πέρας. Εγκρίνεται. 42 δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές ελέγχουμε. πέρας και εγκρίνεται. Είναι κάτι ασαφές. Ψηφίσαμε την 42 δεύτερο τμήμα. Ψηφίσατε σωστά ή όχι. Όχι. Ωραία. Ξαναψηφίζουμε. Αφού δεν κατανοήσατε τι ψηφίζουμε. Λοιπόν, 42 δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Και εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε 46 46 επαναλαμβάνει η πρόεδρος και στα Ιταλικά πέρας εγκρίνεται 47 υπέρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές, τι ψήφισαν οι σοσιαλιστές. Ωραία. Απορρίπτεται 63 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 60. Όχι, επισφύσουμε ψηφίσουμε. Καταπίπτει. Γιατί απορρίφθηκε 63. 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ κατά Αποχές από ε, εγκρίνεται, εγκρίνεται. 69 υπέρ. Α, καταπίπτει. 70. Ωραία, μου δίνετε αντιφατικές γνώμες. Λοιπόν, 69 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 70 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ, κατά, αποχές, λοιπόν, υπέρ, ξανά, κατά, αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 84 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 84 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται ένα υπέρ κατά ε, απορρίπτεται 2 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 6 και 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται 8 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 13 υπέρ, κατά αποχές 13 υπέρ, ξανά, κατά, αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε την 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 18 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 19 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 20 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 23 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ, Θέλετε να λέξουμε την 23. Τι θέλετε, τέλος πάντων. Μα ψηφίσαμε την 22. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά η οποία και αρχίζει. Πέρας και εγκρίνεται. τώρα ψηφίζουμε για τις εγκαταστάσεις στα λιμάνια για την υποδοχή αποβλήτων. Ξεκινάμε με το 1. Τροπολογία 1. Μία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά ελέγχουμε. Τέλος. Απορρίπτεται η 70. Τρία συμβεβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 79. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ, κατά αποχές. Ελέγχουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ κατά α καταπίπτει συγγνώμη 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ. Να ελέγξουμε την 114 υπέρ ήταν οι σοσιαλιστές και το ΕΛΚ. Εννοείται ότι εγκρίθηκε. 118 υπέρ κατά, απορρίπτεται. 119 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 120 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 121 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 122 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 128 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 129 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 131 υπέρ, κατά, αποχές. Δεν βλέπω καλά τα χέρια σας. Επαναλαμβάνουμε, 131 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 33. Τέλος. Απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για το σύνολο του κειμένου. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται. Η επόμενη ψηφοφορία αφορά την κυκλική οικονομία, το διευθυντικό πλαίσιο. Ξεκινάμε με την τροπολογία 8, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 14 αρχή της ψηφοφορίας τέλος εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές από τους σοσιαλιστές είδα μόνο ένα χέρι ελέγχουμε την 19 Τέλος. Απορρίπτεται. Μπορείτε να σκόνετε τα χέρια σας. Σας παρακαλώ. Μπορώ να πηγαίνω λίγο πιο αργά. Λοιπόν, 20 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε την 20. 20. Τέλος. Εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά αποχές ελέγχουμε την 29. Τέλος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 αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ, κατά αποχές. Ελέγχουμε την 43. Τέλος. Εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51 υπέρ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 And now the pie la, la pièce de résistance. Euh, um, Ψηφίζουμε το σχέδιο έκθεση για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας και τροποποίηση της οδηγίας 2011-2024 Ξεκινάμε. Συμβιβαστική 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μ' αρέσει να ακούω σελίδες να γυρίζουν. 57. Υπέρ. Στη σελίδα 10 είμαστε. Νομίζω δηλαδή. Τροπολογία 57. Υπέρ. Κατά έλεγχος. I think it's adopted. The vote is closed. And it is adopted. Compromise 38 in favor. Συμβαστική 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Good work. Πολύ ωραία. Μ' αρέσει. Μ' αρέσουν οι συμβαστικέ τροπολογίε. Compromise 41. Συμβαστική 41. Υπέρ. Στη σελίδα 30 είμαστε. 30. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. to see. um, good. We vote on 41? We voted yes. Yeah, yeah, yeah. Um, I'm trying to see what's happening in the room. Προσπαθώ να δω τι γίνεται στην αίθουσα. Περνάμε στη συμβαστική 42. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 43, στην 435. 35, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Now, uh, IMCO 43. IMCO 43, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έλεγχος, έλεγχος. No. It's closed. Rejected απορρίπτεται. Συμβαστική 44 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Compromise 40. Συμβαστική 45 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 46 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Στη σελίδα 42, συμβαστική 47, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 52. Υπέρ. Κατά. αποχέ Εγκρίνεται. 530. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 54. Υπέρ. Ξέχασα κάτι, λέει πρόεδρος. Όχι. Στην 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. It's rejected, but I, cannot bet on it. The vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. 55. Συμβαστική 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 144. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 161. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήμικο 70. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 595 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Την 7. And it is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχέ. εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. 197 υπέρ, κατά εγκρίνεται. απορρίπτεται.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 Συμβαστική 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήτρε 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά Κυρία Σολατά, γιατί ψηφίζετε κατά. 41 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 241 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 315 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ωραία. 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται. I have never ever seen. Ποτέ μου δεν ξανάδα τόσο καλό αποτέλεσμα. Όλοι συμφωνείτε. Ποτέ δεν ξανάδα τόσες πολλές συμβαστικές. Εγκρίνεται λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια στην κυρία Καβεθόν Ρουίς. Έχουμε μία άποψη της ανεψηφίας, Κυρία Μελά. Oui, merci. Ναι, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να διαβάσω την άποψη της μειοψηφίας. Πρόκειται για μια νομή η οποία είναι επεξήγηση της αρνητικής μας ψήφου, αν υπήρχε μεγάλη ομοφωνία. Όσον αφορά μια κοινή αξιολόγηση αυτών των εχνολογιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαμβάνει κατά την άποψή μας πολλούς κινδύνους. Πρώτον, την αρχή της επικουρικότητας. Σας παρακαλώ πολύ, ακούστε με. Σας ευχαριστώ που με αφήνετε να μιλήσω. Πρόκειται επίση και για μία μαρτυρία εκ μέρους τη Γαλλία. Πρόκειται για κάτι το οποίο ήδη υπήρξε στη χώρα μα. Όταν έγινε η πρώτη εξήμιση των ιατρικών θεραπευτικών αγωγών και των φαρμάκων είδαμε ότι σαν αποτέλεσμα υπήρχε η μη επιστροφή των ποσών με αποτέλεσμα να εξαφανιστούν πολλές ειδικότητε και πολλά εργαστήρια. Το ίδιο θα γίνει και για πολλά φάρμακα στην Ευρώπη, παρόλο που έχουν την πιστοποίηση η Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπουμε ότι πολλές θεραπευτικές αγωγές, πολλές τεχνικές μπορεί να εξαφανιστούν και αυτό το λέει και στο κείμενο βλέπουμε ότι τελικά θα παρεμποδιστεί η δυνατότητα να παρέχεται αυτή η ιατρική περίθαλψη και γι' αυτό και ζητάμε να υπάρξει εδώ προσφυγή στο Συμβούλιο. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας συνεδρίαση. Η επόμενη συνεδρία θα λάβει χώρα στο Στρασβούργο την 1η Οκτωβρίου. Ευχαριστώ πολύ και καλή σας μέρα.